Γενική Ενοχή για τον Ακροτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων από την Επιτροπή Δικαιωματών Γυναικών και Ισότητα των Φίλων. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκαρσία Πέρε, η οποία είναι εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο κριτηρισμός γεννητικών οργάνων των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κορισιών. Ε, ε, μιλάμε για ανισότητα μεταξύ των φύλων και αποτελεί τεράστια εισαγωγή διάκριση κατά των γυναικών. Γίνεται πάντα σε ανήλικέ και αποτελεί επίση παραβίαση και των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίση, παραβιάζει το δικαίωμα στην υγεία, την ασφάλεια και τη σωματική ακαιρεότητα. 140 εκατομμύρια γυναίκε στον κόσμο υποφέρουν αυτή τη στιγμή από τις συνέπειες αυτής της πρακτικής. Δεκεμβρίου του 2014 η Γενική Συνέλευση των Εθνών υιοθέτησε ένα ψήφισμα για να εντατικοποιήσει τι προσπάθειες για την εξάλληψη του κροτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων. Εκεί ζητείται από τα κράτη να αναπτύξουν, να υποστηρίξουν στρατηγικές και τις θέσουν σε εφαρμογή που να απαγορεύουν αυτή την πρακτική επίσης και την κατάρτιση ε, του ιατρικού προσωπικού και των τοπικών και θρησκευτικών ηγετών προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες αρρωγής στις γυναίκες και στα κορίτσια που είναι σε κίνδυνο εδώ σε αυτή τη συζήτηση θα αναφέρω το κάτι άλλο που ανήκει στην Επιτροπή για την καταπολέμηση των ακροτηριασμών γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη μέρα. Εγώ ήμουν 12 ετών και η αδερφή μου 10. Όπως όλα τα καλοκαίρια ήμασταν ε, στο σπίτι ε, των παππούδων μου. Μία μέρα πήγαμε να δούμε τη θεία μου, την αδερφή του πατέρα μου, που πάντα θέλαμε να την επισκεπτόμαστε. Εγώ δεν υποψιζόμουν τίποτα. Η θεία μου με πήγε στο μπάνιο και αυτή και άλλε γυναίκε έπεσαν επάνω μου, με άρπαξαν και μου άνοιξαν τα πόδια. Εγώ ούρλιαζα. Ε, δεν είδα το μαχαίρι, όμως ένιωσα ότι με έκοβαν. Με ραγούσα πολύ, έκλαψα, αλλά μου έλεγαν δεν πρέπει να κλαις. Είναι ντροπή να κλαίει μια γυναίκα. Τώρα είσαι μια γυναίκα. Η μητέρα μας ε, ήρθε να μας δει την πρώτη φορά, έκλαψε και μας φίλησε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στην Αφρική η οικογένεια του πατέρα έχει δικαίωμα ζωής ή θανάτου του παιδιού μα έλεγαν ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι εύρωστη, να είναι συγκρατημένη και να μην μιλάει πολύ. Αυτή είναι μια πραγματική μαρτυρία, όπως εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη συνεχίζουν να είναι θύματα της αδικίας και της ανισότητας στις χώρες της Ένωσης όπου ζουν γυναίκες θύματα αυτή της πρακτικής. Αυτή η πρακτική γίνεται ε, κυρίως κατά τη διάρκεια μιας διαμονής στη χώρα προέλευσης και υπήρχουν και κάποιε ενδείξει ότι γίνεται στην επικράτεια τη Ένωση. Μία μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων Μα έλεγε ότι υπάρχουν θύματα ακροτηρισμού τουλάχιστον σε 13 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2013 δημοσίευσε μια ανακοίνωση με τίτλο Προ την εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, όπου υπάρχει μια εγκάρσια οπτική για την εξάλληψη αυτή τη πρακτική. Γι' αυτό θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συζήτηση για να ρωτήσουμε την Κομισιόν ποιε δράσει έχει αναλάβει στο θέμα αυτό και πώ θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν ειδικού δείκτε να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία και πώς θα συνεισφέρει σε αυτή την πολιτική στις εξωτερικές της σχέσεις. Επίσης, θα θέλαμε να μας πείτε πώς θα εγγυηθείτε η εργασία σας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα της δικαιοσύνης ε, σχετίζεται με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις για να τεθεί τέλος στη βία κατά των γυναικών υπάρχει και άλλη μια ερώτηση στην οποία πρέπει να ευαισθητήσουμε την προσοχή μα και θα ήθελα την απάντησή σα. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εγγυηθεί την προστασία όσων ζητούν άσυλο για θέματα που έχουν να κάνουν με δημοκρατισμό γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο τη οδηγία τη αναθεωρημένη για του ετούντε άσυλο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μα απασχολούν το να μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτή την πρακτική με συγκεκριμένες δράσεις ε, που να είναι της αρμοδιότητάς μας, να εξελίψουμε τον ακροτηρισμό γενικών οργάνων. Πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτό για τη διεθνή στρατηγική. Αν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι αυστηρά, τότε η προσπάθεια θα πάει μάταια. Πρόκειται για μια πρακτική που θίγει τα πιο βασικά δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και έχει πολύ σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες. Όταν μια γυναίκα ενημερώνεται γι' αυτό, ίδια πρέπει να προστατεύσει τις κόρες της και τα άλλα κορίτσια της κοινότητας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το έργο συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων θεσμών και των οργανώσεων που ε, δραστηριοποιούνται στην κοινωνία των πολιτών. Γιατί είναι σημαντικό για να πετύχουμε το στόχο να θεθεί τέλος στην Ευρώπη μια τέτοια ακτινώδης πρακτική που δεν χωρά στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Γιατί αν κάποιο θέλει να αιτιολογήσει αυτή την πρακτική χρησιμοποιώντα κάποιε δικαιολογίε, α πούμε ξεκάθαρα και με δυνατή φωνή ότι σεβασμός στις παραδόσεις και στους πολιτισμούς έχει ως απαραβίαστο όριο το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Περές. Η κυρία Γιουρόβα για την Κομισιόν. Ε, I want to thank... Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την κυρία Γκαρσία Περές για τις προσπάθειες που κάνει για την απάλληψη αυτού του ακροτηριασμού στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 2013 καταγγέλλεται η πρακτική αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει στεναρά τη θέση της κατά όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών ε, συμπεριλαμβανομένου του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των παιδιών. Παραβιάζει την ε, αρτιότητα και σωματική ακαιρεότητα των ε, νεαρών γυναικών ε, επηρεάζει την καλή τους φυσική κατάσταση και υγεία και μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθούν τις δράσεις που αναλάβαμε ε, να προχωρήσουμε στα πλαίσια της δήλωσης. Τι κάνουμε τώρα για την καλύτερη ενημέρωση. Μπορεί να υπάρχουν και 125 εκατομμύρια διεθνώς, όπως δείχνουν οι μελέτες και 500.000 στο... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λίγες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το πώς, από ποιον ε, γίνεται ο ακροτηριασμός αυτός. Η βελτίωση της γνώσης λοιπόν είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θέλουμε να ε, καταρτήσουμε δείκτες και κοινή μεθοδολογία για να υπολογίσουμε τον κίνδυνο του ακροτηριασμού σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Οι μελέτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου θα μας πούν περισσότερα για τους λόγους ε, πίσω από τη συνέχιση ή την εγκατάλειψη του ακροτηριασμού των γυναικείων ε, γεννητικών οργάνων μεταξύ μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταρτήσουμε αποτελεσματική στρατηγική για να τερματιστεί η πρακτική αυτή. Αυτό που κάνουμε τώρα και αυτό που θα κάνουμε στο μέλλον για την πρόληψη τώρα. Για να επιφέρουμε την κοινωνική αλλαγή που χρειάζεται ώστε οι οικογένειες να εγκαταλείψουν την παράδοση αυτή, μόνο η ε, Η νομοθετική δράση δεν αρκεί. Θα πρέπει να ε, έρθουμε σε επαφή με τις κοινότητες που κάνουν τους αγροτηριασμούς αυτούς. Θα πρέπει να τους ενημερώσουμε. Ε, γίνεται λοιπόν προκήρυξη διαγωνισμού για 4,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα ε, διεθνικό πρόγραμμα το οποίο σκοπό έχει να καταπολεμήσει τις ε, επιβλαβείς αυτές επικίνδυνες πρακτικές στην Ένωση. Η Κομισιόν τώρα χρηματοδοτεί τέσσερις ενημερωτικές καμπάνιες που έχουν στόχο συγκεκριμένο τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων. Σε εξωτερικές μας δράσεις επίσης στηρίζουμε ε, βασικά προγράμματα που σκοπό έχουν την αποφυγή αυτού του, αυτής της πρακτικής. Πρόκειται για προγράμματα που εστιάζουν στη δικαιοσύνη, τη δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος για τα δικαιώματα των γυναικών. Χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, μια πλατφόρμα ε, δικτυακή θα ε, καταρτιστεί για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με κοπέλες που διατρέχουν κίνδυνο ή θύματα του ακροτηριασμού αυτού. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια αυτή σήμερα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση που θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών. Πώς προστατεύουμε τα θύματα. Τα... Η οδηγία για τα θύματα θα... το Νοέμβριο του 2015 θα πρέπει να περάσει στις εθνικές νομοθεσίες. Τα θύματα αυτού του ακροτηριασμού θα έχουν έτσι εύκολη πρόσβαση σε καλά ε, δομημένες και λειτουργικές ε, υπηρεσίες που θα, τις, ε, θα τα καλύπτουν κατά τη διάρκεια των δικών και των ανακριτικών διαδικασιών. Υπάρχει συνεννόηση με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή τη οδηγία αυτή, Η τελευταία έγινε 6 Φεβρουαρίου την περασμένη εβδομάδα που ήταν η Διεθνής ημέρα για μηδενική ανοχή κατά του ακροτηριασμού αυτού. Η Κομισιόν επίση διανέμει ενημερωτικό υλικό για τον ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων για τους νομομαθείς ε, μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Τέλος, λίγα λόγια σχετικά με την εξωτερική διάσταση του έργου μας η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η προώθηση της νομοθεσίας ε, για την προστασία των γυναικών συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μην υποφέρουν από παραδοσιακές επιβλαβείς πρακτικές. Ε, όλα αυτά ε, ενσωματώνονται στην πολιτική της Ένωσης και την εξωτερική της δράση για τις γυναίκες. Προώθηση της ισότητας των φύλων. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το, το διάλογο για τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα με όλες τις κυβερνήσεις ε, όπου θέτουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υγείας των γυναικών. Ε, δεύτερον, επίσης ε, είμαστε υπέρ των πρωτοβουλειών ευαισθητοποίησης ε, και την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών για τα δικαιώματα των γυναικών παντού και τρίτον, ε, στηρίζομαι πρωτοβουλίες ε, δημιουργίας ικανοτήτων ε, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Μια φορά το χρόνο γίνεται εκπαίδευση ειδική για το, τη διάσταση του φύλου. Ε, καλύπτει το προσωπικό από την εξωτερική δράση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, γίνεται στα κεντρικά, ε, στις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη-μέλη επίσης. Από το 2012 η Διεθνής Αμνηστία προσεκλήθη να κάνει ε, μία ε, παρουσίαση με θέμα τον τερματισμό του ακροτηριασμού των, ε, του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε με την κυρία Νέγρη από το ΕΛΚ, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας υπέρ της μηδενικής ανοχής στον ακροτηριασμό. Το ΕΛΚ δεσμεύεται στον αγώνα για την εξάλληψη αυτής της τρομακτικής πρακτικής του ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων. Αυτή η υπόθεση πρέπει να τελειώσει παντού στον κόσμο. Εκατομμύρια νεαρές γυναίκες, κορίτσια, υφίστανται αυτό το βασανιστήριο, την, αυτόν τον ακροτηριασμό ο οποίος ε, δημιουργείται, υποτίθεται στο όνομα κάποιας ε, πολιτιστικής παράδοσης ή θρησκευτικής ενδεχομένω παράδοσης. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο 500.000 γυναίκες, νερά κορίτσια εφίστανται αυτήν την απαραίτητη πρακτική. Χαιρετίζουμε λοιπόν ως ΕΛΚ την προσήλωση και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που παρουσιάστηκε ήδη από τον Νοέμβριο του 2013 στην προσπάθειά μας αυτή. Όμως ε, λείπουμε πολύ που δεν έχουν γίνει και πολλά παρά τις φιλόδοξες διακήρυξεις. Τα λόγια δηλαδή δεν ε, συνοδεύτηκαν από πράξεις και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε και τι πετύχαμε στο διάστημα αυτό. Επιπλέον, δεν θεσπίστηκαν συγκεκριμένα πρακτικά αποτελεσματικά μέτρα που θα συμβάλλουν στην εξάλληψη των ακροτηριασμών. Σημαίνω λοιπόν κυρία Επίτροπε τις δηλώσεις σας, τις ανακοινώσεις σας και την δέσμευσή σας υπερμελλοντικών δράσεων. Έτσι πως μας τα είπατε εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου. Τα σημειώνουμε λοιπόν αυτά. Χαιρόμαστε. Αυτό άλλωστε ήταν και ο στόχος της προφορικής ερώτησης. Να πάμε παρακάτω, να κάνουμε κάτι. Από σήμερα λοιπόν έχουμε έναν χάρτη πορείας, αλλά ας μην περιμένουμε και πάλι ένα χρόνο για να κάνουμε κάτι για το θέμα. Θέλουμε οι δεσμεύσεις παρακαλώ να γίνουν πράξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η κυρία Ρένα από τους σοσιαλιστές, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την εισηγησή σας, την περιγραφή των δράσεων που σκοπεύει να λάβει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι, ο κατάλογος είναι πλήρης. Καλύπτει την πρόσβαση στην υγεία, την προστασία των νερών κοριτσιών, των γυναικών, την προστασία των τούντων άσυλο. Χαίρομαι λοιπόν που η Κομισιόν κάτι κάνει για την πρόληψη των ακροτηριασμών. Σύμφωνα όμω με τη συνάδελφο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε με έναν κατάλογο, συμφωνία, αλλά τι γίνεται με τις συγκεκριμένε δράσεις και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το είπατε και εσείς, κύριε Επιτροπή, είναι δύσκολο να συλλέξουμε στοιχεία. Τι γίνεται, θα κάνουμε κάτι προκειμένο. Δεν ξέρουμε επίση τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη, αν έχουν αποτελεσματικέ διαδικασίε και αν υπάρχουν πώ θα τι αξιολογήσουμε. Παρέχεται τη διεθνή προστασία σε αυτά τα νεαρά κορίτσια, τα οποία όμω δεν θα πρέπει να κινδυνεύουν με παραπρόθεση στις χώρες όπου κινδυνεύουν με ακροτηριασμό. Υπάρχουν περιοχές, μάλλον χώρες που απαγορεύουν τον ακροτηριασμό, αλλά υπάρχουν περιοχές σε αυτές τις χώρες όπου η πρακτική συνεχίζεται. Το να στείλουμε λοιπόν πίσω σε μια τέτοια χώρα ένα νερό κορίτσι δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα ίσα Χρειάζεται λοιπόν τα κράτη-μέλη να κάνουν πολύ περισσότερα στον αγώνα κατά των ακροτηριασμών. Καλώ λοιπόν ο κατάλογο καλών προθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένα τι προτείνει το Συμβούλιο για την εφαρμογή στην πράξη αυτού του καταλόγου καλών προθέσεων. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, κύριε Φωνστόρτ, από την ΣΥΑΡ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα του ακροτηριασμού αυτού φαίνεται ότι δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η έννοια θυμίζει τις τελειτουργίες των αφρικανικών φυλών. Και αυτό θα ήταν τρομερό, αλλά τώρα το πρόβλημα έχει μεταναστεύσει σε εμά. Και διαπράτεται εδώ στις χώρες μας επίσης. Είναι ένα φρικαλαίο έγκλημα. Ο ακροτηριασμός των ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν ανήκει στο δικό μας πολιτισμό, δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο δικό μας πολιτισμό. Δεν θα ανεχθούμε τον ακροτηριασμό αυτόν, δεν θα τον αποδεχτούμε. Δεν ακροτηριάζονται σε μας άνθρωποι, ούτε άνδρες, ούτε γυναίκες, ούτε νέοι, ούτε μικρά κορίτσια και μωρά. Τέλος. Ε, σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα στην Αφρική θα ήθελα να πω το εξής. Οι γυναίκες και τα κορίτσια εκεί χρειάζονται βοήθεια είναι 175 εκατομμύρια και κάθε κατέτος προστίθενται 2 εκατομμύρια. Ε, πολλοί, πολλές γυναίκες παίρνουν βοήθεια. Βεβαίως ε, επουδενή όσες θα έπρεπε. Αλλά πάντως ε, υπάρχει κάποια ε, παροχή υπηρεσιών. Και η Ευαγγελική Εκκλησία, η Χριστιανική, δηλαδή οι υπηρεσίες Κάριτας, η Διακονία, η Νίσιο, ε, η Γερμανική Αποστολή, ε, είναι ε, υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια σε αυτά τα κορίτσια. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε το τι παρέχονται τι υπηρεσίες παρέχονται από τις χριστιανικές οργανώσεις. Ε, είναι αναπτυξιακή βοήθεια αυτή που παρέχουν και είναι πολύτιμη η προσφορά τους και στο θέμα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Για την ομάδα των φιλελευθέρων, για δύο λεπτά η κυρία Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ακούτε όσα είπε η Επίτροπος για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράση για την αντιμετώπιση αυτή τη τρομερή μορφή βία κατά των γυναικών και κοριτσιών ακροτηριασμού γενικών γεννητικών οργάνων. Ε, όλοι βλέπουμε τα νούμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακριβώ ε, πόσα κορίτσια ακριβώ υφίσταται αυτή την πρακτική, γιατί δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ε, ε, βάλω τα κορίτσια που συχνά προέρχονται από απομονωμένα τμήματα της κοινότητών μας είναι σε κίνδυνο. Τώρα, πώ θα συλλεχθούν αυτά τα δεδομένα και πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρακτική, αν δεν ξέρουμε το μέγεθο του ζητήματο. Η πρόσφατη ανακοίνωση Κομισιόν δεσμεύεται να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προβούν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των επαγγελματιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη και μοναδική περίπτωση δίκη ε, ε, του γιατρού Νταμαρτσίνα που ε, δεν ε, που δεν συμμετείχε σε κροτηριασμό ήταν ε, μοναδική ότι ποτέ δεν είχε συμμετείχει σε τέτοιες διαδικασίες και ούτε ήξερε κάποια πολιτική των νοσοκομείων. Πρέπει φυσικά ε, να καταρτήσουμε τώρα όλους τους σχετικούς επαγγελματίες έτσι ώστε να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν όταν βλέπουν τις αποδείξεις. Η κατάρτιση παίρνει μόνο κάποιες μέρες αλλά μπορεί να προστατεύσει βάλω τα κορίτσια να αναγκαστούν ε, να ζουν με τι συνέπειε του κριτηριασμού για την υπόλοιπη ζωή του. Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν αρκεί για να τεθεί τέλο σε αυτή την πρακτική. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε στενά με τι κοινότητε, για να αρχίσουν να αλλάζουν οι νοοτροπίε και πρέπει να μιλάμε για το θέμα αυτό, να υποστηρίξουμε τι γενναίες γυναίκες που δεν επιτρέπουν στις, ε, να εκροτηριαστούν οι κόρε του. και επίση θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ε, του κινδύνου και να αντιστεκόμαστε. Σα ευχαριστώ. 1,5 λεπτό για την κυρία Μπιόρκ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ο ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι φρικτό έγκλημα κατά των νέων γυναικών. Η πατριαρχική βία παίρνει πολλές μορφές, αλλά πάντα ο στόχος είναι η καταπίεση των γυναικών, ο περιορισμός του ζωτικού τους χώρου, της σεξουαλικότητας, ο περιορισμός της παρουσίας τους και του ρόλου τους ε, στα δημόσια. Η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών έχει βαθιές ρίζες στις παραδόσεις μας. Ο κροτηριασμό των γεννητικών οργάνων είναι ιδιαίτερα άσχημο παράδειγμα βία κατά των γυναικών. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να εντάξουμε το θέμα αυτό σε πολλά οριζόντια προγράμματα. Πρέπει να ε, φροντίσουμε να ε, ευεργετηθούν από τα προγράμματά μας όλες οι γυναίκες ε, που διατρέχουν κίνδυνο. Θα πρέπει να ταχθούμε κατά της πατριαρχικής βίας της κοινωνίας μας που αν θέλετε μια εκφανσή τους είναι η ατιμορρησία των βιαστών ε, που η απειλή του βιασμού ε, είναι μια συνεχής απειλή ε, η βία αποτελεί έγκλημα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει γρήγορα να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα καταπολεμεί κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών συμπεριλαμβανομένου του ακροτηριασμού. Δύο λεπτά για τον Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Επίτροπο που βρίσκεται εδώ μαζί μας και θέλω και να συγχαρώ την συγκήτρια γιατί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα κατάλληλη ερώτημα. Παρουσία εδώ, αν ε, και είναι μειοψηφική, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρει μόνο τις γυναίκες αυτό το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να ενδιαφέρει όλη την κοινωνία. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που τέθηκε αυτή η ερώτηση γιατί εδώ έχουμε τεράστια απόσταση μεταξύ των λόγων της Κομισιόν και των ε, ε, γεγονότων. Είναι πολύ καλή η ανακοίνωση του Νοεμβρίου 2013, αλλά δεν βρέπουμε να, γίνονται τα κατάλληλα βήματα για να υλοποιηθεί. Θέλουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ο κροτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι ένα έγκλημα που πρέπει να διωχθεί εκεί όπου επιτελείται. Γι' αυτό η Κομισιόν πρέπει να απαιτήσει από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμη δεν εφαρμόζουν την αρχή τη παγκόσμιας δικαιοσύνης να το κάνουν και να διώκουν και αυτούς που οδηγούν τις ε, κοπέλες σε σεξουαλικές χώρες για να τις ακροτηριάσουν, έτσι ώστε να ξέρουν ότι δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Ο ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων που αποτελεί ε, καταρχήν ε, μια βία οπρακία κατά των γυναικών. ουσιαστικά πότε θα αναλάβει δράση η Κομισιόν κατά αυτού, αλλά δεν είναι μόνο νομικό το πρόβλημα. Μόνο 41 περιπτώσει ακροτηριασμού γυναικείων γενικών οργανών έφτασαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ενώ έχουμε 500.000 ε, θύματα. Πολλέ από τι γυναίκε που υφίσταται ούτε καν ξέρουν ότι πρόκειται για έγκλημα και πολλέ άλλε δεν μπορούν ε, να φτάσουν στα δικαστήρια επειδή τι πιέζει η οικογένειά του. Πρέπει να δώσουμε δύναμη στι γυναίκε για να καταγγείλουν, για να ξέρουν ότι όλα τα ευρωπαϊκά όργανα είναι δίπλα του. Πρέπει να εργαστούμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ένταξη, ε, γιατί όπω λέει και η UNICEF, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση είναι τα κλειδιά για να συνεχιστεί αυτή η πρακτική στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ισχυρέ εκστρατείε ευαισθητοποίηση, ε, ανθρωπιστικέ πολιτικέ ασύλου και μετανάστευση. Χρειαζόμαστε ολιστική εστίαση και προσέγγιση που ζήτησε το Κοινοβούλιο και τώρα επαναλαμβάνει. Σα ευχαριστώ λεπτό για την κυρία Μπούρτς ε, για το EFTD. Ε, thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν δεκάδες ε, χιλιάδες περιπτώσεις ακροτηριασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και ούτε ένας δεν προσήχθη στη δικαιοσύνη. αυτή η κατάσταση ε, οφείλεται στην ελευθερία των διαφορετικών ε, εθνοτήτων να ε, συνεχίζουν τα έθιμά τους. Ε, πολλές φορές ε, αντιμετωπίζονται ως ρατσιστές εκείνοι που θέλουν να παρέμβουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δημιουργεί φόβο. Και έτσι συνεχίζονται οι πρακτικές αυτές. Ε, έτσι εγκαταλείπονται οι χιλιάδες ε, ε, γυναίκες και κορίτσια. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αναλάβουμε δράση, να έχουμε το θάρρος. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη, το, την πολιτική ορθότητα που είναι ξεπερασμένη. Κυρία Μπούτσα, υπάρχει μια μπλε κάρτα. Δέχεστε, αν και να, θα περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό μπλε καρτών. Δέχεστε την μπλε κάρτα, παρακαλώ. Uh, e Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να πολεμήσουμε τον κριτισμό γυναικών γεννητικών οργάνων και στην Ευρώπη, αλλά γιατί το UPEN ήθελε να ψηφίσει υπέρ του Ευρωπαϊκού, του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013 που καταδικάζει τον ακροτηριασμό. Νομίζω ότι το UKIP θα ε, πρέπει να βάλει κατά μέρου την αντιευρωπαϊκή ιδεολογία του και να δεχτεί ότι μερικέ φορέ αν εργαστούμε μαζί είναι ο καλύτερο τρόπο για να αλλάξουμε τον κόσμο προ το καλύτερο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν ήμουν εδώ όταν κατατέθηκε αυτό, αλλά οι φιλελεύθεροι έχουν αναλάβει μεγάλη, ε, έχουν πάρει μεγάλη ενοχή στους ώμους τους ε, με αυτή την πολιτική της πολιτικής ορθότητας. Νομίζω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι πραγματικά ντροπή. Η κυρία Μαϊέρ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι αδιανόητο ένα νερό κορίτσι 15 ετών να υφίσταται αυτήν την βία στο πλαίσιο μιας ιασδήποτε τελετής. Πρόκειται για ακροτηριασμό. Τα θέματα είναι 150 εκατομμύρια, μισό εκατομμύριο ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην χώρα μου μόνο έχουμε 28.000 τέτοιες περιπτώσεις ε, εις βάρος γυναικών από τη Σομαλία, την Ερυθρέα, την Αίγυπτο. Απεριγραπτή κατάσταση. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι σε πολιτικό επίπεδο σήμερα για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτών των ακροτηριασμών. Ας μην ε, ξεχνούμε και τον ρόλο του Ισλάμ στο γιατί η γυναίκα είναι σε αυτή τη θέση σήμερα στην Επίρο μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κλείνουμε αυτόν τον γύρο της συζήτησης. Κυρία Στρασφάραχουτ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε από το Λαϊκό Κόμμα καταδικάζουμε την πιο καταφορή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνιστά ο κριτηρισμό γενικών οργάνων. Κάθε 6 λεπτά μια κοπέλα είναι θύμα. 28 χώρες ε, συνεχίζουν ε, να ε, υλοποιούν αυτή την πρακτική. Δεν υπάρχει κανένα θέμα εθήμου ή παράδοση. Είναι βία, είναι έγκλημα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έλεγε ότι πάντοτε είναι μια καλή στιγμή για να κάνουμε το σωστό η Η ε, Ντι Γουαριστήρη, που είναι μοντέλο και ακτιβίστρια, έσπασε τον κώδικα της σιωπής και δείχθηκε στον κόσμο την εμπειρία της όταν ακροτηριάστηκε, ε, όταν ήταν μόνο τριών ετών ε, από μία ηλικιωμένη πραγματικά ήταν ο χειρότερος ακριτηριασμός που μπορούσε να υποστεί μια ηλικιωμενη πραγματικα ηταν ο χειροτερος ακροτηριασμος που εκείνη τη στιγμή διορίστηκε ως εκπρόσωπο του ΙΟΙΕ και ε, ο άνδρας ε, τη μέρα του γάμου του παίρνει ένα μαχαίρι και κροτηριάζει τη γυναίκα του και αν πει το οτιδήποτε τότε εκδιώκεται και τη συμπεριφέρονται σαν να είναι ιερόδουλοι. Ε, μια γυναίκα πρέπει να είναι κροτηριασμένη για να είναι καθαρή και αυτό ουσιαστικά αποτελεί απόδειξη της παρθενίας της. Έτσι λοιπόν ως συνέπεια οι γυναίκες επάσχουν από σωματικές και ψυχολογικές νόσους σε όλη τη ζωή τους. Υπάρχει μια περιμία Σομαλία που λέει ε, ότι η τελευταία καμήλα στην ουρά πάει τόσο γρήγορα όσο η πρώτη. Σίγουρα ό,τι γίνεται στους άλλους και μας μας πλήττει. Γι' αυτό σήμερα ζητάμε από την Κομισιόν κάτι περισσότερο από πολιτική βούληση για να θέσει τέλος στον ακροτηριασμό γυναικών γενικών οργάνων. Θέλουμε πρόληψη πιο αποτελεσματική οικονομική καταστολή από τα κράτη-μέλη, ευαισθητοποίηση, αλλά κυρίως εξάλληψη σε παγκοσμίο επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γουόρτ για ένα λεπτό. Συγκινήθηκα με όσα αγωνίζονται για την καταπολέμηση αυτών των ακροτηριασμών όσων υποστηρίζουν τις γυναίκες θύματα και που προσπαθούν να φέρουν την αλλαγή. Οι εκστρατείε ε, έχουν κάποιο χρόνο ζωή. Τα προβλήματα όμω δεν εξαφανίζονται. Πρέπει να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε μέχρι να πετύχουμε τον τελικό μα στόχο, μηδενική ανοχή. Και ένα καλό τρόπο να το πετύχουμε αυτό είναι να κινητοποιήσουμε τι κοινότητε που θίγονται, να του πούμε τι ιστορίε αυτών που υπήρξαν θύματα ακροτηριασμού, να καταστήσουμε τον ακροτηριασμό στίγμα και να κινητοποιήσουμε και τους γιατρούς, τους λειτουργούς της υγείας, ε, δικαστικούς, ε, νομικούς, δικηγόρους. Πρέπει αυτή η ιστορία να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, πρέπει από οπουδήποτε αλλού. Και πρέπει βεβαίως να συζητήσουμε το θέμα πιο ανοιχτά, να συζητήσουμε το θέμα με διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας διαφορετική γλώσσα, να φτάσει το μήνυμα. Κυρία Ζητνάσκα, ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικά χρόνια διάβασα το ρόδο της ερήμου, ένα βιβλίο το οποίο με βοήθησε να μάθω για την, την πρακτική η οποία επιβιώνει και ακόμη και σήμερα τον ακροτηριασμό των γενικών γεννητικών οργάνων. Υπάρχουν νεαρέ γυναίκε, νεαρά κορίτσια, παιδιά τα οποία εφίστανται αυτό το τρομερό βασανιστήριο και η πρακτική αυτή ε, εννοείται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο πολλά μάλλον ούτε καν για λόγου ε, υγεία γιατί προκαλείται αιμορραγία προκαλείται βλάβε. Ε, ανομαλίες στον εμμινοκύκλο των γυναικών και το καθεξής. Καταδικάζουμε λοιπόν αυτή την πρακτική απερίφραστα. Πρέπει η πρακτική να απαγορευθεί με νόμο σε ορισμένες αφρικανικές χώρες όπως ε, στην Κοντιβουάρ. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ στην Ευρώπη για να προλάβουμε αυτές τις πράξεις τιμωρώντας αυτούς που τις διαπράττουν. Ευχαριστώ. Ο λόγος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιουρεβά. Ο κρατηριασμό γυναικείων κινητικών οργάνων είναι μια ακτινόδη σκληρή και μια ανεκτική πρακτική. Είναι παγκόσμιο έγκλημα κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν ε, δέχομαι δεχόμαστε κάποιος να επικαλείται την ιδιωτική ζωή, τη θρησκεία, τι παραδόσει. Ο κρατηρισμός είναι ένα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ε, τρομοκρατία για να γίνει ε, όπλο πολέμου το σώμα των γυναικών. Ε, Χιλιάδε γυναίκε έχουν κρατηριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω σήμερα να ζητήσω συγκεκριμένα μέτρα να υπάρχει βάση δεδομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένο προπολογισμό και χρονοδιάγραμμα και να επικυρώσει ολοκληρώσει η Ένωση τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, όταν δώσαμε στον γιατρό μου τον, ε, το βραβείο Ζαχάροφ. Πρέπει να θυμηθούμε ότι είπε ότι όταν ακροτηριάζουν μια γυναίκα είναι η γυναίκα μου, η κόρη μου την οποία ακροτηριάζουν. Κυρία Βαλίνα, ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι βέβαιο ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί μία από τι πιο κτηνώδει πρακτικέ και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, στις γυναίκες και στα παιδιά αλλά είναι ε, και η πιο ακραία πράξη πατριαρχικής εξουσίας ε, στο γυναικείο σώμα. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ακροτηριασμό ως μια μορφή δίωξης που βασίζεται στο φύλλο και πρέπει να ακολουθήσουμε τις συστάσεις της ΥΠΑ τη Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών ε, για τις γυναίκες πρόσφυγες. Αν και δύσκολο θα γίνει αυτό, ενώ υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία ε, που προβαίνουν σε επιστροφές θερμό. Ε, και αυτή η πρακτική είναι ένα θέμα που ανησυχεί όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες που πιστεύουν στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και στη δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους. Και εδώ δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ευχαριστώ κύριο Σκοράου. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι και συναδέλφισες, γιατί έχουμε περισσότερες γυναίκες εδώ. Ε, πρόκειται εδώ για μια βαρβαρότητα και ακούστηκε ότι περίπου 3 εκατομμύρια γυναίκες στο χρόνο υφίστανται ακροτηριασμό και περίπου 8.000 στην μέρα. Μιλάμε δηλαδή για 58.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί ακροτηριασμοί γίνονται απευθεία στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Έχουμε διάφορες πρακτικές ε, που έχουν ε, και ψυχολογικές αλλά και σωματικές συνέπειες. Γυναίκες από τις οποίες αφαιρείται ίδια τους η σεξουαλικότητα και η ψυχή. Μιλάμε για βαρβαρότητα. Επομένως, συμφωνώ με την Επίτροπο όταν λέει ότι θα πρέπει να δράσουμε στον τομέα της πρόληψης και το σχέδιο δράσης θα ήταν κάτι καλό, αλλά σίγουρα πρέπει να εργαστούμε και επί του δικαίου του ασύλου σε σχέση με τον επαναπατρισμό των ε, ανθρώπων στις χώρες αυτές. Κύριε Γκουντέφ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πώς να μην είμαι θα υπέρ της μηδενικής ανοχής. Πρόκειται για βάρβαρη πρακτική ενάντια στον πολιτισμό μας και τις αρχές μας. ...500.000 γυναίκες στην Ευρώπη ήδη υφίσταν αυτή την πρακτική... ...λόγω και της μαζικής ε, εισρωής μεταναστών που δεν αφομοιώνονται. Έτσι εγκαθίστανται διαφορετικές πρακτικές στην Ευρώπη. Εσείς είπατε να παράσχουμε προστασία στα θύματα μέσω του ασύλου η επίπτωση αυτού του μέτρου θα ήταν να ενθαρρύνουμε στις χώρες καταγωγής αυτές ακριβώς τις βάρβαρες πρακτικές, δημιουργώντας δηλαδή ένα νέο κανάλι μετανάστευσης. Όχι, πρέπει να ποινικοποιήσουμε τους ακροτηριασμούς, να δημιουργήσουμε έναν κατασταλτικό μηχανισμό και να, μια αρμοδιότητα. Αλλιώς δεν θα υπάρχει καμία προστεμένη αξία στις δράσεις μας. Κύριε Γαμπριέλ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε υπενθυμίζω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία θρησκευτική, κοινωνική, πολιτιστική ή άλλη υπέρ του ακροτηριασμού. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι παίρνει από το χέρι μα, για να τερματιστεί αυτή η πρακτική. Πρόκειται εγκληματική πρακτική. Όσον αφορά την ανακοίνωση τη Κομισιόν του Νευρίου του 2013, συμφωνούμε εννοείται όλοι. Είναι πιστική ανάγκη. Χρειάζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να θέσουμε τέρμα στην πρακτική αυτή. Επιμένω επίση στον ρόλο κλειδί που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φίλων. Πρέπει να θεσπίσουμε συγκεκριμένου δείκτε για να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Τρίτον, όσον αφορά την εξωτερική πτυχή, την πολιτική κρίζωση αυτή τη πρακτική, ευθύνω την προσοχή σα στην σημασία συνεκτική στάση και συντονισμού μεταξύ ημών, κυρία Επίτροπε, και όλων των φορέων που υπερμείνονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρακολουθούν την μετανάστευση. Συντονισμό, ανταλλαγή στοιχείων, συμπληρωματικότητα λοιπόν. Αυτέ είναι οι τρεις λέξεις κλειδί. Τέταρτον, να αναστοχαστούμε το πώ συνδέονται οι ακροτηριασμοί με την πολιτική μετανάστευση. Το άσυλο δεν είναι λύση. Συν υπάρχει πάντα ο τα κορίτσια αυτά να επαναπροωθούν στις χώρες καταγωγής. Επίσης όχι στο επιχείρημα της ε, προστασίας της υγείας. Πρόκειται για έγκλημα. Και ας κοιτάξουμε εν τέλει να μην ε, αντικαταστήσουμε ένα λάθος με ένα χειρότερο. Κύριε Ροντρίκης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ το θέμα αυτό για το ακροτηριασμό ε, δεν έχει να κάνει με την θρησκεία, με την παράδοση. Είναι έγκλημα. Εκατομμύρια γυναίκες έχουν ακροτηριαστεί. Επίσης, 200.000 βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν έχουμε νόμους που να ογκιώνται την ασφάλεια των γενικών σε Ευρωπαϊκή επικράτεια δεν τρέχουν κίνδυνο του ακροτηριασμού. Ακόμη στην Ευρώπη έχουμε μεσαιωνικά έθιμα ο κρατηριασμό γυναικείων κινητικών οργάνων είναι ένα από αυτού. Δηλαδή έχουμε μια βάρβαρη, απαθή Ευρώπη μπροστά σε κάποια νούμερα που ούτε καν μπορεί να επιβεβαιώσει. Η κυρία Επίτροπος λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα στατιστικά στοιχεία. Όμω είτε ήταν 50 είτε 500 χιλιάδες γυναίκες. Ε, ε, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Όλοι εξογυρώμαστε με τα νούμερα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ε, Όμω, θα συνεχίζουν αυτά τα μαχαίρια να κόβουν τις γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν λάβει συγκεκριμένα μέτρα και αν δεν εμπλακεί σοβαρά δεν θα πατήχουμε τίποτα. Ευχαριστώ κυρία Βιτσινιέσκα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, παρακολουθώ προσεκτικά τη συζήτηση και είμαι ε, εξοργισμένη. Ε, εννιά φορές γιορτάσαμε το έτος μηδενικής ανοχής στον ακροτηριασμό. Και τι γίνεται. 140.000 στον κόσμο ακροτηριάζονται. 2 εκατομμύρια το χρόνο είναι τα θύματα. 500.000 ε, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τρομακτικά στοιχεία που έχουμε σήμερα τον 21ο αιώνα σαδιστικά ε, ε, έθιμα μπορεί να μιλάμε και να συζητάμε αλλά στην πράξη πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες ποιος θα βοηθήσει αυτές τις γυναίκες αν όχι εμείς σήμερα κυρία Επίτροπε τι συγκεκριμένα μέτρα προτείνετε κυρία Φορέντσα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συναδέλφοι, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ε, τη συζήτηση μας να την βάλουμε στο σωστό πλαίσιο. Το θέμα δεν ε, είναι η ε, χριστιανική ποιότητα της Ευρώπης, ούτε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο δρόμο εκτοξεύοντα ρατσιστικά συνθήματα όπως άκουσα. Αν εμείς θέτουμε την αυτοδιάθεση των γυναικών, της ελευθερία των γυναικών και το παραβίαστο του σώματος του στη βάση των ε, ιδεών μας. να εμείς ακούσουμε ε, την επιτακτική ανάγκη να σταματήσουμε την άσκηση βίας ε, των ανδρών επί των γυναικών. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε Ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε να περιμένουμε να ε, υπογράψει τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λείπουν στατιστικά στοιχεία, ο Eurostat ε, που δίνει στατιστικά στοιχεία για, το για όλα τα πράγματα δεν ξέρει ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος στην Ευρώπη. Μία μέρα όπως ε, σήμερα όπου θρυνούμε και άλλα θύματα στη Μεσόγειο Ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας. Διακόπτει την ομιλήτρια Πρόεδρος, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, κυρία Επίτροπε, και πριν από ένα χρόνο ε, είχατε μιλήσει για την ανακοίνωση αυτή. Πέρασε ένας χρόνος, όμως η πρακτική αυτή πλήττει εκατομμύρια. Είναι καταχρηστική πρακτική ε, και όχι μόνο, είναι έγκλημα και θα πρέπει να υπάρξουν νόμοι που θα ποινικοποιούν την, ε, τον ακροτηριασμό. Θα πρέπει να καταδικάζονται και οι ένοχοι γονείς ε, και όλοι όσοι ε, διαπράττουν το έγκλημα αυτό. Θα πρέπει να σταματήσει η ατιμορρησία. Επίσης έχουμε ευθύνη και μέσα από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, δηλαδή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση για τα δικαιώματα των παιδιών και τους ιατρικούς κινδύνους αυτών αυτής της βάρβαρης πρακτικής που προκαλεί σωματική και ψυχολογική ζημιά στα κορίτσια. Πρέπει να στηρίξουμε τις τολμηρές θαραλές γυναίκες που τολμούν να καταγγείλουν αυτά όπως στην Σενεγάλη ε, που υπάρχει μη κυβερνητική οργάνωση που ενισχύει τις γυναίκες αυτές ε, να καταπολεμήσουν το, τη βαρβαρότητα. Θα πρέπει να σεβαστούμε βεβαίως ε, ξένους πολιτισμούς και παραδόσεις. Όχι όμως να δεχτούμε τη βία κατά των παιδιών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι νομιμοποιείται από το διαφορετικό πολιτισμό ή την παράδοση ή το έθιμο. Παρακαλώ λοιπόν να ανταποκριθείτε στο καλό σας όνομα και αναλάβετε δράση. Ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Νίλσεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μία παράδοση χιλιετής ε, οι κοινωνίες εξυγχρονίζονται αλλά η πραγματικότητα του ακροτηριασμού παραμένει για εκατομμύρια ε, ανθρώπους, γυναίκες και θεωρείται ο ακροτηριασμός ταμπού στις χώρες ε, και περιοχές όπου ασκείται. Ε, δεν είναι μόνο ένα σωματικό πρόβλημα, είναι, είναι κάτι περισσότερο, σαν να σου το στόμα ε, ίσως. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να χαράξουμε μια πολιτική για τις γυναίκες ε, που θα είναι οριζόντια σε όλους τους τομείς και θα να ε, συνεχίσουμε να εργαζόμεθα μαζί με τις γυναίκες σε συνεργασία μαζί τους σε όλο τον κόσμο. Κυρία Γκέρλινγκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Όλοι συμφωνούμε εδώ ότι ο ακροτηριασμός είναι από τις πιο βάρβαρες μορφές ε, προσβολής της σεξουαλικότητας των γυναικών και της ζωής τους ολόκληρης. Το θέμα σήμερα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη εμείς Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο το γεγονός ότι ε, όλοι εδώ έχουμε καθίσει για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ε, οι διώξει είναι πολύ χαμηλές. Πρέπει να ε, αναδείξουμε βέλτιστες πρακτικές, να εξασφαλίσουμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη ε, να ε, φροντίσουμε για την επιτυχία των πολιτικών μας. Ακούσαμε να γίνεται λόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις τελευταίες προσπάθειες ή τις πρώτες προσπάθειες για διώξεις. Ε, ο Πρωθυπουργό πριν από ένα χρόνο ε, διέθεσε ε, ένα σημαντικό ποσό περίπου 4 εκατομμύρια στερλίνες για να γίνει πολιτική κατά των ακροτηριασμών. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η ενημερωτική εκστρατεία και να διευρυνθεί παντού. Ο πρωτηριασμός γυναικείων γενετικών οργάνων ε, είναι μία από τις πιο κατάφορε πρακτικές βία κατά των γυναικών. Παραβιάζει τα δικαιώματά τους αλλά και τα δικαιώματα των παιδιών και ε, προκαλεί τεράστιε ζημίες ε, στην ψυχολογία, στο σώμα τους και πολλές φορές φτάνει και στο θάνατο. Είναι η πιο κτηνώδης μορφή άσκηση βίας από τα πατριαρχικά συστήματα και μάλιστα ακόμη παραμένει αόρατη. περισσότερα πέρα από, τα, πέρα πλαίσιο δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την πρακτική πέρα από χωρίς να ενισχύσουμε τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, χωρίς να βελτιώσουμε την υγεία των παιδιών και της μητέρας. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά θίγονται από το μακροκομμενικό μακροοικονομικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τι συμβαίνει ε, στις χώρες μας και πρέπει να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα που έχουν και οι γυναίκες αυτές. Η κυρία Ματέρα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Το 2006 το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά ε, έθεσε αυτό το θέμα του ακροτηριασμού ε, και ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί εκτάκτως ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το φαινόμενο, αν και συμβαδίζει με πολύ διαφορετικές κουλτούρες από τις δικές μας, ε, πολλές γυναίκες ε, υφίστανται αυτή την πρακτική και ζουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Νοέμβριο του 2013 ο θεσμός που εκπροσωπείται ανέλαβε μια σειρά δράσεων για την καταπολέμηση αυτού του βάρβαρου φαινομένου, όμως η έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος καθιστά πολύπλοκη τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την πραγματική αποτελεσματικότητά του. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη στο να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία που να εμποδίζουν αυτή την πρακτική να συνοδευτεί και με πραγματική βοήθεια στα θύματα. Θα πρέπει να εργαστούμε για να υποστηρίξουμε την κοινότητα και τους επαγγελματίες του κλάδου αυτού. Το Φεβρουάριο γιορτάσαμε τη Διεθνή ημέρα κατά το κριτηρισμό Γενικών γυναικείων γεννητικών οργάνων. Αν ε, θέλουμε να έχει συγκεκριμένη σημασία η μέρα αυτή και αν θέλουμε να συνεισφέρουμε στην εξάλληψη του φαινομένου, θα πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Σας ευχαριστώ, Κύριο Μαρτών, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Διπιστώνω ότι λίγοι άνδρες μίλησαν για την μάστιγα αυτή και είναι κρίμα. Ας αφήσουμε τα στερεότυπα. Το θέμα αφορά και τους άντρες, αφορά την ανθρωπότητα ολόκληρη. Το πρόβλημα είναι ο ακροτηριασμός, ο ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων. Ακροτηριάζουμε γυναίκες, τις τραυματίζουμε, πολλές φορές βρίσκουν το θάνατο. Πρόκειται για αποτέλεσμα μιας βαθιά ριζωμένης ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το είπατε άλλωστε, δεν είναι αφρικανικό μόνο το πρόβλημα, αφορά και την Ευρώπη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να προαγάγουμε την αλλαγή της νοοτροπίας. Και βεβαίω να επικυρώσουμε την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεδομένου ακριβώ ε, του προβλήματος, της μάστιγας αυτής. Οι γυναίκες αυτές δεν μπορούν να είναι θύματα. Πρέπει να είναι μαχητές, όπως έλεγε και ένας γνωστός ε, γιατρός. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε. Κύριε Βεσέλη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μία εικόνα αξίζει χίλιες φορές, μάλλον πολύ περισσότερο από χίλια λόγια. Εγώ ε, είδα την εικόνα μιας γυναίκας ε, που έχω τη φωτογραφία μιας γυναίκας που κρατά ε, το μαχαίρι γιατί το να προβαίνει κάποιο σε σκόπιμο ακροτηρισμό γυναικών γενικών οργάνων είναι έγκλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αναγνωρίζουν πώς περπατούν οι γυναίκες που έχουν ακροτηριαστεί, πώς μπορεί να εξετάρει κάποιον κάτι που προκαλείται από τον πόνο. Αυτό οδηγεί στο να εργαστούν οι γυναίκες ε, για να βρουν σύζυγο. Ε, τώρα εδώ έχω μια μαρτυρία. Εγώ ήμουν 9 ε, χρονών, μου είπε ο πατέρα μου να ανέβω στο αυτοκίνητο ότι θα πάμε σε μια γιορτή. Δεν ήρθαν τα αδέρφια μου, θυμάμαι μόνο μια γυναίκα με ένα μαχαίρι και τον πατέρα μου που με κρατούσε από τον μπράτσο. Αυτό έγινε στην Ισπανία το 1993, όμως περισσότεροι κροτριασμοί γίνονται στις χώρες προέλευσης η Ισπανία έχει ένα πρωτόκολλο ε, που δεσμεύει τους γονείς να μην ακροτηριάζουν τις ε, κόρες τους. Νομίζω ότι αυτό το πρωτόκολλο θα έπρεπε να υιοθετηθεί σε όλη την Ένωση. Χρειαζόμαστε επιγόντως νομοθετικά και χρηματοοικονομικά μέσα για να προστατεύσουμε τα θύματα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε διάφορα πιστεύω, να κάνουμε ό,τι υπάρχει στο χέρι μας, ό,τι είναι στο χέρι μας για να θάψουμε αυτό το μαχαίρι που ακροτηριάζει το σώμα και την ψυχή των κορτσιών. Κύριε Πλυνκεβιτσιούτε, κύριε Πρόεδρε, οι ακροτηριασμοί αυτοί εις βάρος κοριτσιών είναι βαθιά ριζωμένη πρακτική σε πολλές περιοχές του κόσμου. Είναι πιο βάρβαρη μορφή διάκρισης κατά των γυναικών. Είναι μια μορφή, μια ακραία μορφή ανισότητας που σου δυστυχώς και στην Ευρώπη. Απειλεί την υγεία, τη σωματική ακαιρεότητα των γυναικών, οι οποίε δεν είναι δυνατόν να βασανίζονται σήμερα το 2015. Δεκάδε χιλιάδες γυναίκες στην Ευρώπη κινδυνεύουν από τέτοιου είδους ακροτηριασμό. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ισότητας των Φίλων... μόνο 41 υποθέσεις έφτασαν στα δικαστήρια. Τι κάνουμε λοιπόν για την βία αυτή κατά των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει την πράξη διατάξει για να τιμωρηθούν αυτοί που είναι ποινικά υπεύθυνοι. Κύριε Επίτροπε, περιμένω από εσά συγκεκριμένη δράση. Κύριε Κύριε Πρόεδρε, περίπου 140 εκατομμύρια νεαρές γυναίκες σε όλο τον πλανήτη υφίστανται ακροτηριασμό των γενετικών τους οργάνων. 150.000 στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται ότι οι λόγοι είναι πολιτιστικοί. Αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό το επιχείρημα αυτό όταν θίγονται βασικά θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Ο ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων πλήττει την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν είναι δυνατόν να υφίστανται οι γυναίκες αυτές βασανιστήρια. Ιδιαίτερα σήμερα. Είναι παραβίαση του δικαιώματο στη ζωή. Από το οποίο απορρέουν και όλα τα άλλα δικαιώματα. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες. Πρέπει να αγωνιστούμε για να εξαλείψουμε αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές. Αυτοί οι ακροτηριασμοί διαπράττονται σε πάνω από 20 χώρες της ε, Αφρικής, σε χώρες που ενισχύουμε με αναπτυξιακή βοήθεια. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε την βοήθεια αυτή ως εργαλείο πίεσης για να βελτιώσουμε βεβαίω την κατάσταση και όσον αφορά τι παραβιάσει και άλλων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν και τον Επιτρόπο Μίτσα, σκοπεύει να κάνει κάτι προ την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντα αυτά τα εργαλεία. Ευχαριστώ. Κύριε Τζουφρίντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πριν λίγες μέρες, την Παγκόσμια ημέρα, ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεία διέδωσε τεράστια νούμερα αυτής της σκληρής πρακτικής. Υπολογίζεται ότι έχουμε 830.000 κορίτσια σε κάποιες χώρες όπως την Αίγυπτο, στη Γουινέα, περίπου το 90% του γυναικείου πληθυσμού υφίστανται αυτή την πρακτική. Όμως και στην Ευρώπη, στην Ιταλία, Ιταλία μας λένε ότι τουλάχιστον 40.000 γυναίκες ε, υφίσταται αυτή την ε, σκληρή πρακτική που τις ε, καθιστά αντικείμενο. Ε, πρέπει να αγωνιστούμε για μια νομοθεσία που να απαγορεύει αυτή την πρακτική και να προβλέπει κυρώσεις και να παρέχουμε κατάλληλη βοήθεια στα θύματα, να προωθήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης ε, για να εξαλειφθεί μια τέτοια πρακτική. παραπέμπουμε στην έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας και δίνουμε κουράγιο και στις γυναίκες θύματα. Ευχαριστώ κυρία Ρέγκνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πολλοί από εμά αποστήλαμε το ίδιο μήνυμα. Όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούμε. Όλοι οι βουλευτές λέμε ότι ο ακροτηριασμός των γεννητικών γυναικείων οργάνων ε, συνιστά αδίκημα και το συμπέρασμα είναι κοινό ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα πλαίσια δεν πρέπει να συζητεί αλλά να δρά. Αναφέρθηκαν οι ενημερωτικές εκστρατείες, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, να αναλάβουμε δράση και να φροντίσουμε να συνιστά λόγο παροχής ασύλου ο ακροτηριασμός. Εμείς οι Ευρωπαίοι ε, βουλευτές πρέπει να ταχθούμε υπέρ αυτής της λύσης με όσο γίνεται περισσότερες φωνές. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε στο τμήμα ΚΑΤΣΔΙ. Ένα λεπτό, κυρία Πίτιερ. Ευχαριστώ. Ο ακροτηριασμός γενικών γεννητικών ε, οργάνων ε, πολύ νεαρών κοριτσιών προκαλεί πολύ σοβαρές συνέπειες και πάρα πολύ μεγάλο πόνο, μολύνσεις, επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και στη γέννα συχνά οδηγεί σε θανάτους. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις συνέπειες ε, αυτής της απάνθρωπης πράξης. Ο κροτηριασμός παραβιάζει σοβαρά την αξιοπρέπεια των γυναικών και των κοριτσιών παγκοσμίω και παραβιάζει και τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών. Τα κορίτσια συχνά κροτηριάζονται και στην Ευρώπη ή τα πηγαίνουν στη χώρα προέλευσης των γονιών τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα κορίτσια δεν θα γίνονται θύματα και θα πρέπει οι γονείς τους να τιμωρούνται για μια τέτοια πράξη. Κυρίως Σερασάντος, ε, για γενικά θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο δράση ε, και για το μέτρο που ανακοίνωσε. Είναι σχεδόν απίστευτο ότι πρέπει να μιλάμε για αυτό το θέμα στον 21ο αιώνα. Και μάλιστα ρωτιόμαστε πώς φτάσαμε ω εδώ, πώ είναι δυνατόν μία τόσο κτηνώδη πρακτική να λαμβάνει χώρα στον κόσμο μα και μάλιστα στην Ευρώπη, στη χώρα μου. Έχουμε ε, κάποιες περιπτώσεις, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ε, σε όλη την Ευρώπη όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν φτάνουν. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε να υπάρχει μια προσπάθεια που να στοχεύει στην εκπαίδευση, να υπάρχουν εκπαιδευτικές εξτρετίες για τις κοινότητες που υπάρχει μεγαλύτερος κινδύνος να συμβεί αυτή η πρακτική. Η Κομισιόν θέλει να λάβει έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της άσκησης βίας κατά των γυναικών και θα πρέπει να υπάρχει και εφαρμογή της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Κύριος Μαριάς. Η έκθεση που συνέταξε το 2013 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων η σύγχρονη αυτή βαρβαρότητα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Η έκθεση διαπιστώνει ότι υπάρχουν θύματα ή δυνητικά θύματα σε τουλάχιστον 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η δυνητικα θυματα σε τουλαχιστον 13 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξυ των οποιων η γερμανια στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ω εκ τούτου ο κίνδυνο υποβολή στην πρακτική αυτή θα πρέπει να αποτελεί βάσιμο λόγο για τη χορήγηση ασύλου ή ανθρωπιστική προστασία. Τέλο, για την εξάλληψη του ακροτηριασμού θα απαιτηθεί σειρά ενεργειών που επικεντρώνονται στη συλλογή δεδομένων στην πρόληψη στην προστασία των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο στην ποινική δίωξη των δραστών και την παροχή υπηρεσιών για τα θύματα. ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ο είναι κοινό. Ακούμε τρομερά πράγματα απόψε και λυπάμαι πραγματικά που η παρουσία των βουλευτών είναι πολύ περιορισμένη. Είμαστε κανένα τριραριά εδώ, τη στιγμή που υποφέρουν εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Κρίμα που υπάρχουν μάλιστα και τόσο λίγοι άνδρες Και οι γυναίκες, ξέρετε, έχουν δικαίωμα σε σεξουαλική ζωή. Γι' αυτές δίνουμε μάχη. Ο αγώνας θα είναι μακρύς βεβαίως. Πρέπει να πείσουμε όλους τους άνδρες του πλανήτη να συμμετάσχουν στον αγώνα αυτόν. Γιατί καλό είναι να λένε οι πολιτικές ομάδες ότι πρέπει να αγωνιστούμε, αλλά μένουν να γίνουν πολλά για να εξελίψουμε αυτό το απότροπο φαινόμενο. Κύριε Ζεπόσκα. Κύριε Πρόεδρε. Οι ακροτηριασμοί αυτή είναι μια απίστευτη πρακτική όσο και να σέβουμε τις θρησκευτικές πεπιθήσεις ή ουδήποτε αλλά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η βαρβαρότητα στο πλαίσιο οποιασδήποτε θρησκείας. Το φαινόμενο έχει καταδικαστεί πολλάκις ε, η δική μας συζήτηση δεν πηγαίνει όμως ε, δυστυχώς αρκετά μπροστά. Δηλαδή, το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πράξη με τον πιο χειρό, με τον πιο έντονο τρόπο, με συγκεκριμένα μέτρα. Φοβούμε όμως ότι δεν είναι θέμα της Ευρώπης ναι κυρώσει τη συμβέρεση τη Κωνσταντινούπολη. Είναι θέμα των κρατών μελών. Κύριε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ω άνθρωπο και ω γιατρό, βρίσκω αποτρόπαιη την πρακτική. Πρέπει να λάβουμε μέτρα αμέσως, χωρίς την παραμετρή καθυστέρηση. Να διώξουμε τους υπευθύνους ακόμη και εξοδαφικά. Μισό εκατομμύριο θύματα ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως ακούσαμε 41 μόνο υποθέσεις ήρθαν ενώπιον των δικαστηρίων. Ντροπή. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για ένα πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζουμε παρκώς. Πρέπει να διευνήσουμε αυτήν την πρακτική και να ενημερώσουμε, να προετοιμάσουμε τους λειτουργούς της υγείας. Να προστατεύσουμε αυτούς που θίγονται άμεσα, αυτούς που κινδυνεύουν. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν έδωσε η Κομισιόν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρά μόνο ένα ευχολόγιο. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την υιοθέτηση αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για να τελειώσει αυτή η νοσηρή πρακτική στο έδαφος της Ένωσης. Όμως θα έχουμε πρόβλημα και με την καλύτερη νομοθεσία. Το, το πρόβλημα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας. Χρειάζεται μεγάλη αποφασιστικότητα από τα κράτη-μέλη που μέχρι τώρα δεν πέτυχαν να τερματίσουν αυτές τις πρακτικές στο έδαφος τους ως μέρος μιας πολιτικής δημόσιας υγείας αυτό δεν πρέπει να είναι μεμονωμένο μέτρο, πρέπει να είναι ευρύτερα ενσωματωμένο στις κοινωνίες μας. Η απομόνωση αυτών των κοινοτήτων τις πρόχνει συχνά στις παλιές παραδόσεις, στις παλιάς τους πατρίδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τραβήξει μια γραμμή εδώ και να πει σαφώς ότι παρά την πολυπολιτισμικότητα αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Διακοπή κυρία Παραντίκα. Ευχαριστώ αυτό το πρόβλημα πρέπει να έχει μια πολυτομιακή απάντηση σε εκπαιδευτικό επίπεδο, υγειονομικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε να πάρουμε καλή δέσμευση και κατάρτιση των κλιματιών γιατί έχουμε μια απάνθρωπη και κτηνόδη υπερακτική που διατηρείται λόγω ε, της έλλειψης ενημέρωσης. Έχουμε υποχρέωση ε, όλοι όσοι πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν να βία δικαιώματα. Πρέπει να αναλάβουμε συντονισμένη δράση για να εντοπίσουμε τον κίνδυνο, να πείσουμε τις οικογένειες ε, που μπορεί κάποιες διακοπές ε, ε, στη χώρα προέλευσης να τις μετατρέψουν σε φιάλτη για τις ε, κόρες τους. Πρέπει να παρέχουμε και ψυχική βοήθεια στα θύματα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και σε τοπικό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε και ευρωπαϊκή στήριξη για τις παγκοσμίες δράσεις. Κύριε Επίτροπε, εσείς ποια στήριξη βρίσκεται στο Σώμα των Επιτρόπων. Ευχαριστώ κύριε Κινίτσι. Ευχαριστώ τα στοιχεία για ε, την πρακτική του κριτηριασμού είναι ενισχυτικά και στις τρίτες χώρες ε, και στην Ένωση και φυσικά είναι μερικά αυτά δεδομένα και έτσι καθίσταται πολύ πιο δύσκολη η στρατηγική πρόληψη και οι στοχευμένε δράσει για τα θύματα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά καταγγελία από τι γυναίκε και για τι ανήλικε. Υπάρχει και κίνδυνο δευτερογενού θυματοποίηση ε, από του γονεί. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικό τα όσα μας παρουσίασε η Επίτροπος, όμως πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες νομοθεσίες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ε, να υπάρχει και πολιτιστική πρόοδος εντός και εκτός Ευρώπης για να αντιμετωπίσουμε και να προκαταλάβουμε αυτή αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή βίας κατά γυναικών και κοριτσιών. Και θα κλείσουμε το Κατσιδιάι με την κυρία Χάνιμπολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο ως κάποιος που εκπροσωπεί μια εκλογική περιφέρεια με κοινότητες όπου γίνονται, γίνονται αυτοί οι ακροτηριασμοί. Είναι βάρβαρο, συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Όμως ε, η επιβολή του νόμου δεν έχει επιτυχία. Δεν έγιναν επιτυχείς διώξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο παρόλο που έχει ποινικοποιηθεί εδώ και καιρό ο ακροτηριασμός. Η Γαλλία ήταν λίγο πιο... τα κατάφερε κάπως καλύτερα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις ίδιες τις κοινότητες να καταλάβουν ότι αυτή η πρακτική είναι λανθασμένη να καταλάβουν, με, ε, να καταλάβουν ε, τις γυναίκες αυτές ε, και πρέπει να στηρίξουμε τις γυναίκες που είναι διατεθειμένες να μιλήσουν κατά του εθήμου αυτού. Αυτό θα βοηθούσε πραγματικά. Ολοκληρώνεται εδώ το ΚΑΤΣΔΙΑΙ και δίνω το λόγο στην κυρία Γιούροβα. Κυρίες και κύριοι, ε, πιστεύω ότι θέλω να σας πω ότι και εγώ είμαι σοκαρισμένη από το γεγονός ότι εξακολουθεί να ελοποιείται η πρακτική αυτή και έχουμε και μάλιστα τόσο ψηλά νούμερα και όχι μόνο εκτός αλλά και εντός Ευρώπης. Έχω δει αυτά τα νούμερα πρόσφατα, αλλά πριν από αυτό δεν γνώριζα ότι αυτή η βάρβαρη πρακτική είναι τόσο βαθιά ριζωμένη σε αυτή την Ήπειρο. Εγώ εξέτασα όλα τα διαθέσιμα μέσα στην Ευρώπη αλλά και στα κράτη-μέλη και μπορώ να πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν μια νομοθεσία που καθιστά δυνατή τη δίωξη αυτής της πρακτικής ακόμη και αν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στον ποινικό κώδικα ε, ο κροτηριασμός των γυναικείων κινητικών οργάνων πάντοτε μπορεί να βρει κανείς χα, ε, χάρη ε, να χρησιμοποιήσει την βαριά σωματική βλάβη. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους νομικές δυνατότητες. μιλάμε για μηδενική ανοχή απέναντι στον ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ενώ όταν μιλάμε για μηδενική ανοχή απέναντι στο έγκλημα, αυτό είναι κάτι που το θεωρούμε δεδομένο, κάτι που ούτε καν τίθεται προς συζήτηση. Και όταν ε, μιλάμε για τον κριτηριασμό πολλές φορές, ε, παρουσιάζονται κάποια επιχειρήματα, βλέπετε αυτό είναι παράδοση, είναι κάτι που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και δεν μπορεί να εξαλειφθεί εν μία νυχτή. Εγώ πάντοτε θα υποστήριζα τη διατήρηση των παραδόσεων, όμω μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο για μια παράδοση που πραγματικά καταπατά όλε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε μέσα, όπως παραδείγματος χάρη την νομοθεσία για το άσυλο, Βάσει αυτής της νομοθεσίας, ε, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να προσδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευπαθή άτομα, ιδιαίτερα στις γυναίκες και στα κορίτσια, που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε κίνδυνο να είναι θύματα αυτής της πρακτικής. Έχουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε. Στη συζήτηση αυτή υπόθηκε ότι η Κομισιόν δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει επίση τα κράτη-μέλη. Βεβαίω όχι, αλλά έχουμε το δικαίωμα να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να μην χρονοτριβούν ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας και της καταπολέμησης αυτής της πρακτικής. Αλλά φυσικό είναι δύσκολο να καταπολεμήσει κανείς ένα τέτοιο φαινόμενο αν δεν γνωρίζει ποιο είναι το εύρος του ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Ε, κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουμε λάβει ε, από τα κράτη-μέλη μας δείχνουν ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, όμως από ορισμένα κράτη τα τελευταία στοιχεία που έχουμε σχετικά είναι από το 2007. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πάντοτε καινούργια στοιχεία. Δεν προσπαθούν όλα τα κράτη-μέλη να χαρτογραφήσουν την κατάσταση και πολλά από αυτά τα νούμερα είναι απλές εκτιμήσεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα. Θα έπρεπε λοιπόν να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Στο παρελθόν είχαμε αναφέρει και τη στρατηγική για τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών που καταρτίζουμε. Και ένα σημαντικό σκέλο αυτή τη στρατηγική θα είναι και η καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και εδώ θα αναπτύξουμε ένα σχέδιο δράση και ελπίζουμε ότι αυτό θα μα βοηθήσει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα βήματα. Σύμφωνα όμως με τη δική μου εμπειρία, ένα σχέδιο δράσης δεν θα είναι επαρκιά αξιόπιστο αν δεν έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας και αυτό κάνουμε. Αυτά ήθελα να πω εγώ αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι θα επενερχόμαστε τακτικά στο θέμα αυτό, γιατί είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Πάντοτε θα είμαι στη διάθεσή σας, όχι μόνο εδώ στην Ολομέλεια, αλλά σε διαρκή βάση θα μπορώ να σας ενημερώνω για το τι κάνει η Κομισιόν. Καταλαβαίνω ότι καλείται για την ανάληψη συγκεκριμένων βημάτων και δράσεων και σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση.